Uh, uh, and gentlemen, uh, once again. Κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας, της ΙΤΡΑ. Έχουμε την ε, ημερήσια διάταξή μας που είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Αν δεν υπάρχουν σχόλια μπορούμε να την εγκρίνουμε χωρίς αλλαγές, δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια. Ε, κάτι πολύ σημαντικό που έχω να πω. Η ε, συνεδρίαση για τις, 11, για τις 11 Μαΐου ακυρώνεται. Δεν θα γίνει η συνεδρίασή μας τότε, αλλά θα γίνει η συνεδρίαση στο Στρασβούργο, όπως είπα πιο πριν, την 5η 18 Μαΐου, 9 με 10 και μισή. Ήταν αδύνατο να συμφωνήσουμε με τους δύο εισηγητές και τις δύο επιτροπές ε, σε άλλη ημερομηνία, οπότε 5η 18 Μαΐου ε, στο Στρασβούργο 9 με 10 και μισή. Επόμενη συνεδρίαση της ΣΥΤΡΑ θα γίνει στις Βρυξέλλες την Δευτέρα 29 και 3η 30 Μαΐου. Οπότε, σε τέσσερις εβδομάδες περίπου θα έχουμε την, ε, την ψηφοφορία στο Στρασβούργο για τις πλατφόρμες, για τις ε, επιγραμμικές πλατφόρμες. Τώρα, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, 4, 25-26 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2017. Πρακτικά των δύο αυτών συνεδριάσεων. Έχετε τα πρακτικά στους φακέλους σας. Σημείο 5. Copyright και σχετικά δικαιώματα εφαρμοστέα για ε, συγκεκριμένες ε, επιγραμμικές ε, διαβιβάσεις. Η συγκήτρια η κυρία Μλίναρ δεν είναι εδώ. Αλλά η κυρία Βίρινγκ θα την αντικαταστήσει. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την εισηγήτρια. Να σας θυμίσω ότι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για το φάκελο αυτό είναι η Γιούρη. Η Ήτρε θα υποβάλει την νομοδότησή της επί, του κανόνα, επί του κανόνα 53 ε, και ο προτινόμενος κανονισμός αποτελεί κομμάτι του πακέτου για το copyright με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε περισσότερα α, ε, ε, ραδιοτηλεπτικά προγράμματα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε, να ξεκινήσουμε με την εισηγήτρια, με, τις τα σχόλια της εισηγήτριας από την κυρία Βίρνικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το, μέρος, ε, παίρνω το λόγο συγγνώμη εκ μέρους της ε, Αγγέλικα Μίναρτ. Η εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη οι κανόνε, οι τρέχοντε κανόνε για το copyright να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή. Ως προς αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό που ε, διευρύνει κάποιες αρχές ε, από, για την, από την οδηγία για την καλωδιακή και, την, ε, και τις τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου για τους, για, που μπορεί να παραταθεί για τους παρόχους ραδιοτηλεπτικού περιεχομένου. Η η συγκήτρια στηρίζει την γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αφορά την επέκταση της αρχής της χώρας καταγωγής των ραδιοτηλεπτικών παρόχων και την διεύνηση των, της διαχείρισης συνολικών δικαιωμάτων για τις υπηρεσίες της ραδιοτηλεπτικές. Σε ό,τι αφορά την αρχή της χώρας προέλευσης, η συγκήτρια πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βρει την ε, ισορροπία μεταξύ των ε, κατόχων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ε, πρόσβασης στις ραδιοτηλεπτικές στο περιεχόμενο. Ε, επίσης ε, περιλαμβάνονται ε, υπηρεσίες που δεν είναι ε, παραπλευρές ό,τι αφορά τις μεταδόσεις και η ε, προσέγγιση της ε, Κομισιόν επιτρέπει στην αγορά να, προσαρμόσει την, ε, να προσαρμοστεί στις, αγορές, στις αλλαγές και τις νομικές επίσης τροποποίησεις. Η πρόταση δεν έχει στόχο να υποβιβάσει τον, το, την, την, γεωγραφικούς περιορισμούς ή την ελευθερία των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαριστούν τα όσα έχουν να κάνουν με, την, με τον ανταγωνισμό και να γίνει μια αναθεώρηση του αντικτύπου αυτού του κανονισμού. Κυρίως ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τις ε, επενδύσεις στα ραδιοτηλεπτικά ε, έργα μόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Ό,τι αφορά την παράταση την, ε, της διαχείρισης συνολικών δικαιωμάτων, η συγγήτρια πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτή μόνο στα κλειστά δίκτυα, αλλά και στις αναμεταδόσεις μέσω του ίντερνετ. Εφόσον ε, υπάρχουν σύνδεσμοι με το, με το περι... ορισμένο ελεγχόμενο περιεχόμενο ε, και μέσω των εγγεγραμμένων χρηστών. Ε, τέλος, η εισηγήτρια υποστηρίζει τα όσα υπάρχουν σε κάποια κρατημέλη όπως η αδειοδότηση. Ε, η συγκετρια βεβαίως προσβλέπει στην συμβολή και στη συνεργασία όλων των συναδέλφων και των ε, σκιωδών συγκητών για την ε, έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε την άποψη της συζυγήτριας. Πάμε στους σκιώδεις. Ο κύριος Σαλίνη, εκ μέρους του ΕΠΠ που αντικαθιστά τον κύριο Πατριτσέλο. Πολύ περίπλοκα αυτά τα πράγματα. Ε, ναι, είμαι κι εγώ ένα αντικαταστάτη τελευταία στιγμή. Οπότε, όπως και συνάδελφος, θα διαβάσω την παρέμβαση του κυρίου Παντριτσέλο που είναι ο Σκιώδης για το θέμα για το οποίο συζητάμε. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια Μίλνερ για τις ε, τροπολογίες που κατέθεσε και που είναι στην ίδια γραμμή με το αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Ο οπτικοακουστικός τομέας της Ευρώπης αντιπροσωπεύει σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της Υπήρου μας με πάνω από ένα εκατομμύριο απασχολούμενους από τους οποίους και με 100 δισεκατομμύρια

Ε, κέρδη ετησίω. Το τομέας της παραγωγής και της διανομής ε, θέλει να έχει εγγυημένη την αποκλειστικότητα του περιεχομένου και της ε, εδαφικότητα. Είναι σημαντικό να μπορούν να τοποθετηθούν στην αγορά και να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Ενώ λοιπόν συμμεριζόμαστε την επιθυμία της Κομισιόν για τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, δεν μπορούμε να μιλάμε υπόψη την ανάγκη για να εγγυηθούμε την ισορροπία ενώ ταυτόχρονα την ανάγκη να προστατεύσουμε επαρκώς τα πνευματικά δικαιώματα των φορέων του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. Το πρότυπο που υπάρχει για την δαφική άδεια έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις που γίνονται σε ψηφιακό περιεχόμενο και για να προστατεύσουν την πολιτιστική διαφοροποίηση των προϊόντων, καθώς και για να ικανοποιήσουν την ανάγκη των καταναλωτών για λογικές τιμές. Η ιδέα της ε, επέκτασης της αρχής της ε, χώρας προέλευσης και για τις ε, υπόλοιπες υπηρεσίες μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λεπτή ισορροπία που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής και που επιτρέπει σε πολλούς φορείς να είναι στην αγορά με βάση τη βασική, το βασικό κανένα της, των πνευματικών δικαιωμάτων που χορηγείται σε κάθε, στη χώρα μάλλον του κάθε δημιουργού. Μπορεί όμως να μην έχουν οι διάφοροι φορείς τη δυνατότητα να πάρουν πανευρωπαϊκές άδειε και γι' αυτό πολλοί μικρομεσαίοι μπορεί να βρεθούν εκτός αυτού του κομματιού της αγοράς. Ταυτόχρονα πολλή παραγωγή περιεχομένου ενώπιον μιας ακατάλληλης προστασίας του δεν θα μειώσουν το περιεχόμενο που μπαίνει στην αγορά, πράγμα που σημαίνει απώλεια για άνω των 8 δις ευρώ ε, σύμφωνα με υπολογισμούς. Η αρχή της χώρας προέλευσης λοιπόν για τις υπηρεσίες online μπορεί ε, να είναι λάθος που θα θέσει σε κίνδυνο τον οπτικοακουστικό τομέα που είναι τόσο σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το φως αυτών των παρατηρήσεων. Είναι βέβαιο ότι χάρη στη συζήτηση και χάρη στις, στις ε, προτάσεις εφαρμογής που θα υποβάλουν και οι άλλοι συνάδελφοι και οι τροπολογίες που θα υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, θα μπορέσουμε στο τέλος των διαπραγματεύσεων να φτάσουμε σε μια γνωμοδότηση με την οποία να συμφωνούμε και να είναι και ταυτόχρονα αρκετά φιλόδοξη, ώστε να δώσει χρήσιμες ε, λαβές και στην Νομική Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε τη γνώμη του σε συγγετή και τώρα θα περάσουμε στον εκπρόσωπο των σοσιαλιστών, τον κύριο Μπλανκολόπεθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το οπτικοακουστικό μοντέλο βασίζεται σε δύο στοιχεία, την πώληση του περιεχομένου σε εδαφική βάση και την αποκλειστικότητα. Το να επεκταθεί η αρχή της χώρας προέλευσης για διάφορες ε, ε, υπηρεσίες ε, online μπορεί να υποσκάψει την αρχή της εδαφικότητας. Εξάλλου, δε, μέσω μπορεί να οδηγηθεί στην απαγόρευση των ε, συμβάσεων ε, κατά αποκλειστικότητα ε, για τις τηλεοράσεις επιπληρωμή. Γι' αυτό μπορεί να βλάψουμε ολόκληρο τομέα. Η πρόταση κανονισμού είναι αδύναμη. Σύμφωνα με την Κομισιόν, βασικός στόχος είναι να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών, γιατί λέει η διαδικασία μέχρι σήμερα είναι περίπλοκη και οι φορείς φέρουν μεγάλο κόστος. Όμως η Κομισιόν δέχεται ότι δεν έχει συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με το κόστος. Υποψιάζομαι ότι η Κομισιόν βασίζει την πρότασή της σε μια ανάγκη που δεν μπορεί να την στηρίξει με στοιχεία. Ε, άρα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής ε, μιλά για βοηθητικές υπηρεσίες, αλλά δεν μπορεί να μας ε, πει τι είναι αυτές οι υπηρεσίες. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, γίνεται λόγος για πολιτιστικά προγράμματα, πολιτικά προγράμματα ή ντοκιμαντέρ, αλλά τίποτα από αυτά δεν ε, περιλαμβάνεται στο διατακτικό. Όσον αφορά τη συμβατική ελευθερία, μιλάμε για αυτή την αρχή σε ένα εκτιμώντας. Ε, δεν κατοχυρώνεται στο διατακτικό και πάλι. Μιλάμε λοιπόν ε, για έναν κανονισμό που όσον αφορά το τμήμα της αναμετάδοσης δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι ε, προσφέρει λύσεις. Οι εμπορικέ τηλεοράσει είναι κατά. Η παραγωγή οπτικοακουστικού ε, περιεχομένου επίσης και οι διανομή αυτού του περιεχομένου επίσης. Οπότε τελικά μόνο γινούνται αμφιβολίες, αν όχι και καθαρή αντιπαράθεση. Ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε βαθιά αλλαγή του πρόταση αυτή σε κανονισμό. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ε, και να ε, καθιερώσουμε την ελευθερία ε, σύμβασης ε, για τους φορείς. Δεν μπορούμε επίσης να αποκλείσουμε αυτές τις υπηρεσίες online που έχουν στόχο κρατήριο εκτός ε, του κράτους μέλους της καθίδρυσης της κάθε εταιρεία. Εάν η Κομισιόν θέλει να αλλάξει το μοντέλο, θα έπρεπε να μας έχει στείλει μια ανακοίνωση για τις προθέσεις της και για τις προθέσεις νομοθετικών αλλαγών, γιατί διαφορετικά δημιουργείται αβεβαιότητα και ανασφάλεια σε αυτό το τομέα που το 2014 ε, ε, παρήγε 86 δις ευρώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εγώ εδώ αντικαθιστώ τον σκιώδη συγκητή μας. Γενικώ συμφωνούμε με τα συμπεράσματα και με την θέση που εξέφρασε προηγουμένως η εισηγήτρια εδώ. Έχουμε δύο διατάξεις, μάλλον δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να ε, θα, θέλαμε. Πρώτον, να μην θίγονται ρυθμίσεις στις χώρες μέλη για δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις ε, συλλογικές συμβάσεις. Και δεύτερο, οποιασδήποτε διαφορές όσον αφορά την άσκηση δικαιωμάτων θα είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας των χωρών μελών. Αυτά θέλουμε. Άλλος κανείς επιθυμεί να λάβει το λόγο, λέει ο πρόεδρος ε, Μπούζεκ όχι. Άρα, ο, προ, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, DG Connect της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, μάλλον συγγνώμη, πρόκειται για κυρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Εγώ αντικαθιστώ τον ε, ε, συναδελφό μου που είναι πραγματιματάρχης και λέγομαι Γιούκνερ, πρόεδρος Μπούζεκ. Τι ωραία, βεβαίω εδώ όλοι δικαστούμε ε, πολύ συχνά άλλου συναδέλφου, έτσι λοιπόν και εσείς. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στο γιατί κατατέθηκε η πρόταση και να εξηγήσω τον στόχο της πριν να έρθω και σε ορισμένε από τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει τα μέλη σας στην σημερινή συνάντηση. Και πρώτα για την ανάγκη που έχετε να καλύψει η πρόταση, δηλαδή για τις ανάγκες των Ευρωπαίων, ότι δηλαδή κάτι έχουμε να τους προσφέρουμε το θετικό. Εδώ για την επιγραμμική τηλεόραση βλέπουμε ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση σχετικά. 42% των Ευρωπαίων ε, παρακολουθούν επιγραμμική τηλεόραση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Υπάρχει και μάλιστα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τέτοιο περιεχόμενο και από άλλες χώρες μέλη. Έρευνα που έγινε προδιετίας έδειξε ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους θέλουν να βλέπουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο από άλλες χώρες μέλη, εκτός της δικής τους δηλαδή. Η ανάλυση που κάναμε για τη μελέτη επιπτώσεων αλλά και η συνεχιζόμενη εργασία μας δείχνει ότι υπάρχει πολύ γεωγραφικός αποκλεισμός και για προγράμματα όπως πολιτιστικά προγράμματα, ντοκιμαντέρ, ε, ψυχαγωγίας, παίγνια, ακόμα και ιστορικά και άλλα σχετικά. Και πολύ σημαντικό δηλαδή πολιτιστικό περιεχόμενο το οποίο ε, αποκλείεται γεωγραφικά. Γίνεται δηλαδή αντικείμενο geoblocking. Στην πρόταση της ε, Επιτροπής στόχος είναι να καταστεί δυνατό στους Ευρωπαίους broadcasters και σε αυτούς οι οποίοι ε, διαχειρίζονται τις επιγραμμικές ε, εκπομπές να έχουν την ευκαιρία να δίνουν περισσότερο, να δείχνουν μάλλον περισσότερο από αυτό το περιεχόμενο στους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι επιγραμμικοί broadcasters, το προτινόμενο μέτρο, θεσπίζει την αρχή της χώρας προελεύσεως που ανοίγει δυνατότητες. Είναι δηλαδή enabling, προσφέρει δυνατότητα, δεν τους υποχρεώνει, δεν υποχρεώνει τους broadcasters, δηλαδή τους σταθμούς και άλλους να εκπέμπουν και πέραν των συνόρων. Ούτε μειώνει την ελευθερία, τη σημαντική ελευθερία να κάνουν γεωγραφική κατανομή, βεβαίω θα πρέπει να σέβονται του κανόνε που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρηκα που άκουσα ότι η συγκέντρια και ορισμένοι από τα μέλη σα υποστηρίζουν τι γενικέ γραμμέ των προτάσεων τη Κομισιόν. Άκουσα βέβαια να εκφράζονται και κάποιε ανησυχίε και θα ήθελα πολύ σύντομα να έρθω στι ανησυχίε αυτέ. Όπω είπα πριν, η πρόταση δεν ανατρέπει το σύστημα χορηγήσεων αδειών στην Ένωση. Σέβεται τα υπάρχοντα και περιλαμβάνει και ορισμένε ε, ρήτρε διαφύλαξη. Δηλαδή, εφόσον τα συστήματα αυτά δηλαδή δεν έρχονται σε αντίθεση με τους υφιστάμενους κανόνες και, και προβλέπεται και αμοιβή για τους ε, αυτούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές προσφέρονται περισσότερα κίνητρα ωστόσο για να χορηγηθούν, να γίνει δηλαδή διαθέσιμο περισσότερο περιεχόμενο διασυνοριακά, προσφέροντας έτσι συγκεκριμένα ωφέλη στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Πολύ σύντομα, διότι άκουσα να μιλούν κάποιοι για την έρευνα για τον ανταγωνισμό. Λίγα λόγια εδώ. Επειδή συνεχίζεται βεβαίως η εκδίκαση υποθέσεως αυτής, δεν πρόκειται να την σχολιάσω, αλλά να σας πω λίγο το ε, νομικό ιστορικό. Κάτι που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι οι αποφάσεις του δικαίου ανταγωνισμού είναι πάντοτε ειδικέ κατά το χαρακτήρα και κατά την υπόθεση και στοχεύουν να αποφευθεί η στρέβλωση ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν όμως γενική εφαρμογή όπως άλλα νομοθετικά εργαλεία. Το ίδιο στο άνθρωπο που μιλούμε και εδώ μιλούμε για συμφωνίες που απαγορεύουν τον ανταγωνισμό. Αυτά έχουν και εξαιρέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, αντιλαμβάνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να έχουν ως αντικείμενο την αποκομίση κέρδους και ιδίως στην διευκόλυνση για το λανσάρισμα νέων προϊόντων. Όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, τα πράγματα δεν είναι ή άσπρα ή μαύρα. Δεν υπάρχει τίποτε στην ε, συνθήκη που να αποτρέπει ή που να απαγορεύει την πρόθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στην κοινή αγορά. Όπως είπα, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε κίνητρα και να επιτρέψουμε να κυκλοφορήσει περισσότερο περιεχόμενο μέσα στη, διαδικτυακό περιεχόμενο μέσα στην Ευρώπη και αναμένουμε τη συζήτηση που θα διεξαχθεί και στην Επιτροπή σας αλλά και ε, μεταξύ ημών και του Συμβουλίου για να επιτευχθεί ο στόχος που προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Βεβαίως, εξ ονόματο τη κυρία Λίνερ. Όχι, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι 27 Απριλίου. 14 στην Ήτρε. 31 Ιουλίου και το Σεπτέμβριο στην Επιτροπή, ε, στην ε, Συναρμόδια Επιτροπή. Άρα η γνωμοδότησή μας θα πρέπει να είναι έτοιμη τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, για τη συνεργασία σας. Το επόμενο θέμα είναι το υπαριθμό 6. Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έχουμε εισηγητή τον κύριο Ζανονάτο. Το μέτρο αυτό είναι μέτρο που εντάσσεται στο πακέτο καθαρής ενέργειας, θα το θυμάστε αυτό. Εδώ έχουμε τρεις σημαντικούς στόχους ενώπιον μας. Κοινή μεθοδολογία για την αντιμετώπιση σενάριων κρίσεων, διαρκή παρακολούθηση της ε, ζήτησης και της ε, παροχής και σχέδια για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρίσεων. Και θα πρέπει να διασυνδέσουμε την νομοθετική πρόταση με τα άλλα τμήματα της δέσμης και ιδίως την ρύθμιση περιπεκτικού ρεύματος, γιατί αυτά συνδέονται πολύ στενά. Τώρα το λόγο έχει ο συγητής μας κύριος Ζανονάτο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κατημέλη στην προετοιμασία και διαχείριση των ε, ενεργειακών κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, ε, ορίζει μάλιστα την κρίση ηλεκτρισμού ως μια σημαντική έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας ή την αδυναμία παροχής ηλεκτρισμού στους τελικούς καταναλωτές. Μιλάμε για ε, γεγονότα τα οποία είναι σχετικά σπάνια, τα οποία όμως για τα οποία ακόμα δεν έχουμε αρκετή εμπειρία διαχείρισης και που μπορεί να έχουν όμως ε, ε, απτό αντίκτυπο και κάποιες φορές και δραματικό αντίκτυπο στις ε, περιφέρειες που πλήττονται. Παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2008 400.000 ήταν οι πολίτες στην βορειοδυτική Πολωνία που λόγω έλλειψη ηλεκτρισμού έμειναν για 18 ώρες χωρίς ηλεκτρισμό. Τον Ιανουάριο του 2009 οι ε, αντίξωες συνθήκε συνθήκες στην Γαλλία οδήγησαν στη διακοπή παροχής ηλεκτρισμού σε 1.250.000 ε, Γάλλους πολίτες. Στην Κύπρο του Ιούλιο του 2011 συνέβη κάτι παρόμοιο, όπως και στη Μάλτα και στη Σικελία τον Αύγουστο του 2014, στη Βόρεια Ορλανδία το Μάρτιο του 2015, για να μην μιλήσουμε για την κρίση λιγρισμού του Ιανουαρίου 2017, δηλαδή πριν λίγους μήνες, στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη και αυτές οι κρίσεις ε, προκάλεσαν ε, ζημιές ε, σημαντικές στις οικονομίες αλλά και πολλές δυσκολίες συχνά δραματικού τύπου στους πληθυσμούς. Είναι καλό να παρατηρήσουμε ότι αυτό το θέμα μας στιγμής έχει αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό πλαίσιο. Και λέω αμέσω ότι αυτή είναι μια πιθανή λύση, αλλά που ως αίτιο έχει προφανή έλλειψη των εθνικών εγκαταστάσεων. Θέλουμε να συνεργαστούμε λοιπόν, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κενό αριθμιστικό που προτείνει να καλύψει αυτή η πρόταση κανονισμού. Το σχέδιο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε τέσσερα άξονες αξιολόγηση του κινδύνου με πρόταση ε, μεθοδολογίας για να εντοπιστούν σενάρια κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο και ε, τα σενάρια κρίσης σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και τη μεθοδολογία για να δούμε πόσο είναι κατάλληλες οι εγκαταστάσεις καθώς και ε, είναι οι αρχές που διέπουν ε, αυτές τις διαδικασίες. Έχουμε διαχείριση κρίσεων, δηλαδή ε, συναγερμός και η επιβολή κατάστασης κρίσης ε, στην αγορά. Τέλος, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση, η ex post. Η δε αυτή παρακολούθηση θα γίνεται από την ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια. Δεν θα μακρηγορήσω για όλες τις τυχές πρώτα, δεν έχουμε το χρόνο και ε, πάντως γενικά είναι ισορροπημένο αυτό το κείμενο και συνδέεται με σημαντικά κεφάλαια του χειμερινού πακέτου για την ενέργεια. Τα επιχειρησιακά περιφερειακά κέντρα που προβλέπονται από τον κανονισμό ΆΣΕΡ στην οδηγία ανανεώσιμες και τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση καθώς και την οδηγία για τη διαχείριση της αγοράς, καθώς και η οδηγία για τη διαχείριση κρίσεων, ε, δηλαδή τον οδηγό, την οδηγία για το, το κανονισμό, με συγχωρείτε, για το άσερα και ε, για τη ρύθμιση της αγοράς. Θα πρέπει ωστόσο να εντοπιστούν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, οικονομική, πολιτική, ε, διοικητική και τεχνική, που αποτελούν εμπόδιο για την προετοιμασία της διαχείρισης των κινδύνων. Και άρα πρώτον, οι πολύ περιορισμένους κρίσεις των διασυνδέσεων ε, σε ένα πλαίσιο που πολλοί φορεί κινούνται με βάση λογικέ προστατευτισμού ως προς την ενέργεια. Έπειτα υπάρχει ένα κενό νομικό όσον αφορά τις μορφές ε, αποζημίωσης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν επίσης τα κράτη-μέλη να πρέπει να είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν ενέργεια προς τα άλλα σε περίπτωση έλλειψης. Άρα λοιπόν από εδώ ξεκινάμε για να δούμε κατά πόσο τα όσα προτείνει η Κομισιόν ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Κυρίως σημαίνει η ανάγκη ε, να υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύστημα αξιολόγησης, προετοιμασίας ε, και διαχείρισης ε, των κινδύνων που να είναι εύχριστο και ευέλικτο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ανάλογα με τις διάφορες πραγματικότητες και σύμφωνα με τα σχέδια της προστασίας ε, των καταναλωτών και της ασφάλειας της ενέργειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, on behalf of EPP. Ο κύριος Νίδερμαϊερ τώρα, εξ ονόματος του έλκα, που είναι ισχυώδης εισηγητής. Uh, <clears throat> Ευχαριστώ. Μιλούμε για αυτό το φάκελο και πρώτα Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο τομέας της ενέργειας και κυρίως του, του ηλεκτρισμού έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Εμείς εισαγάγουμε νέες τεχνολογίες και βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη μας τους στόχους για το κλίμα. Θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτηση από, τις, από τον άνθρακα. Αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις ε, που συνδέονται με αυτές τις νέες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται μία εκ των οποίων είναι η λειτουργία της παραγωγής ε, ηλεκτρικού ε, ε, ρεύματος και η παροχή της, και η σταθερότητα της παροχής. Έχουμε λοιπόν πολλές προκλήσεις, πολλά νέα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, αλλά και νέες ευκαιρίες σε αυτό το πακέτο όπου προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε φτηνή, βιώσιμη και ασφαλή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μικρό το τμήμα αυτό του αφορά τον ηλεκτρισμό, σε ό,τι αφορά το γενικό πακέτο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ε, και κυρίως ό,τι αφορά την ε, αντιμετώπιση, την προετοιμασία για τους κινδύνους και την ε, ασφάλεια της παροχής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι νέες ε, ε, τεχνολογίες ε, με τι προκλήσει που δημιουργούν θα μπορέσουν να... οι προκλήσεις που δημιουργούν μάλλον οι νέε τεχνολογίε θα μπορέσουν να λυθούν. Θέλουμε λοιπόν μια σωστή προσέγγιση ω προ αυτό και αυτό περί αυτού πρόκειται σε αυτό τον φάκελο. Και επίση θέλουμε να έχουμε μια νέα μεθοδολογία έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αναγνώριση των διαφόρων επικίνδυνων παραγόντων. Καλωσορίζω λοιπόν αυτό το κείμενο, αυτή την έκθεση. Είναι πολύ αξιόλογο κομμάτι του συνολικού πακέτου. Ε, μέχρι στιγμής νομίζω ότι είναι κάποια ίσονα σημασία θέματα που παραμένουν εκκρεμή, τεχνικά κυρίω και βεβαίω θα τα συζητήσουμε, αλλά ε, θα ήθελα ο εισηγητή να οργανώσει μια τέτοια τεχνική συνάντηση και να μα ξεκαθαρίσει κάποια διάφορα, κάποιες, ε, ε, θέματα σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες στις διάφορες αγορές, αλλά και κάποια νομικά ζητήματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και θα καταφέρουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι του εξίσου σημαντικού πακέτου να περάσει. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Άλντε, ο κύριος Πέτελσεν που αντικαθιστά την κυρία Μλίναρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους εκ μέρου τη κυρία Μλινάρ να πω το εξή. Καλωσορίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτού του νέου κανόνε για την αντιμετώπιση και την προετοιμασία για του κινδύνου στον ε, τομέα του ηλεκτρισμού και την βελτίωση τη ε, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και διαφάνεια, που είναι βεβαίω σημαντική για την αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και σημαντικό βήμα για να δημιουργηθεί μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση. Η δουλειά που συνεχίζεται σε ό,τι αφορά του κανόνε για τι επίγουσε καταστάσει στον τομέα του αερίου και τη ε, ηλεκτρική ενέργεια δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωση τη νομοθεσία έτσι ώστε να εγγυηθούμε τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού συστήματο και στον τομέα του ηλεκτρισμού. Ε, πιστεύω ότι μια προσέγγιση με βάση την αγορά είναι καλύτερη και σε καιρούς κρίσης. Παρ' όλα αυτά η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε ότι ο ηλεκτρισμός θα φτάνει εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα βήμα προ σωστή κατεύθυνση, καθορίζοντα μια κοινή μεθοδολογία, εναρμονίζοντα ε, τα διάφορα εθνικά σχέδια αντιμετώπιση ε, επικίνδυνων καταστάσεων και βελτιώνοντα την ανταλλαγή πληροφοριών σε ε, περιφερειακό επίπεδο. Αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Κυρίω σε ό,τι αφορά το συντονισμό και την αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που πρέπει να λάβουν υπόψη τι διαφορέ που υπάρχουν στα διάφορα εθνικά συστήματα ηλεκτρική ενέργεια. Τέλο, να τονίσω ότι δεν είναι αρκετό να συντονιζόμαστε μόνο σε περιφερειακό επίπεδο και να βελτιώνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Αν θέλουμε να αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανεπαρκείς ε, συνθήκες σε ό,τι αφορά την αγορά ενέργειας, όπως ας πούμε οι ανεπαρκείς διασυνδέσεις. Οπότε είναι σημαντικό αυτή η πρόταση να, να είναι συνδυασμένη με όλες τις άλλες προτάσεις που υπάρχουν για το καθαρό πακέτο ε, και να περάσει βεβαίως ε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε συνδυασμό με τη δουλειά που έχει γίνει σε όλες, τα, σε όλα τα, όλες τις προτάσεις. Και βεβαίως θα συνεργαστούμε στενά, με τους εισηγητές για να γίνει αυτό ο κύριος Μπενίτο Ζιλουάγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ θετικό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έχει υποβάλει αυτή την νομοθετική πρόταση γιατί για πρώτη φορά έχουμε κάποιες κανόνες που βλέπουν που προβλέπουν μάλλον τις περιπτώσεις έλλειψης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι σημαντικοί αυτοί οι κανόνες, καταρχάς λόγω της αρχής της και δεύτερον για να εγγυηθούμε την παροχή ε, των βασικών και την κάλυψη των βασικών αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών. Ω προ αυτό θα πιστεύω πως θα ήταν καλή ιδέα να αναφέρουμε ποιοι θα είναι και ποιε θα είναι οι βασικές, ε, μάλλον οι πελάτες προτεραιότητες αυτοί που οπωσδήποτε πρέπει δηλαδή να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Δεύτερον πιστεύω ότι στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λείπει η αναφορά στην ενεργειακή επάρκεια ως το καλύτερο δρόμο για την εξασφάλιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μην φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις κινδύνου. Ξέρουμε πως ήδη το έχει κάνει αυτό η Κομισιόν για την παροχή φυσικού αερίου. Επίσης πιστεύω ότι ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε και την αυτοκατανάλωση ε, ως έναν από τους τρόπους για να μειωθεί αυτό το, αυτός ο κίνδυνος. Έτσι θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε και χρήματα για τους πολίτες ε, όσον αφορά το κόστος των υποδομών, υποδομών που πολλές φορές ε, ε, έχουν και αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς και δυσκολίες γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια πάντοτε. Επίσης, αποτελούσε μια καλή όθηση για την ε, ενεργειακή μετάβαση προς ε, πιο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πιο αποκεντρωμένες και πιο ε, δημοκρατικές. Εν γέννη, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι πολύ λεπτομερές όσον αφορά τα προβλεπόμενα μέτρα και αυτό θα πρέπει, μπορεί να οφείλεται στο ότι είναι απλώς ένα σχέδιο ή γιατί μπορεί έτσι να θέλουμε να ενισχύσουμε τις αρχές του enjoy που ε, πρόσφατα έχει δημιουργηθεί. Πάντως, αν η ιδέα είναι οι ιδιωτικέ εταιρείε να συντάσσουν τα σχέδια επίγουσες ανάγκη χωρίς κανένα περιθώριο και χωρίς καμιά σαφή ιδέα, φυσικά είμαστε τελείω αντίθετοι. Η τελική νομοθεσία θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη για το ποια θα είναι αυτά τα σχέδια επίγουσες ανάγκης και να μην αφήσουμε στα χέρια των λόμπι αυτό το θέμα. Να μην δώσουμε δηλαδή στα λόμπι την νομοθετική εξουσία. Ευχαριστώ. Fox, Από όσο βλέπω, ο κ. Χένκελ είναι εδώ και είναι έτοιμος να αντικαταστήσει τον ε, σκιώδη του ECR που λείπει. This was a misunderstanding. I wanted to talk... Παρεξήγηση έγινε, πρόεδρε. Εγώ ήθελα να μιλήσω για το Acer. raise your hand because replacement is quite typical. Εδώ πέρα έχουμε πολλές φορές ε, αντικαταστάσεις ε, στην, ομάδα, στην Επιτροπή μας και νόμιζα ότι θέλατε να μιλήσετε γι' αυτό. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εισηγησή του. Η πρόταση τη Κομισιόν προσφέρει πιο ευρωπαϊκή εστίαση στη προσέγγιση αυτού του θέματο, του συστήματο του ηλεκτρικού. Ε, βλέπουμε ότι προωθείται η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και καλύτερη ε, επίση ε, μείωση της, του κόστου του συστήματο, έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστο κατανάλωση για τον τελικό χρήστη. Το χειμερινό πακέτο το οποίο θεσπίζει ένα ηλεκτρικό σύστημα όπως ας πούμε διαχείριση της ζήτησης, η καλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί συντονισμό ε, όμως πιστεύω πως αυτή την πρόταση εναρμόνισης είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη την ε, διαφορετικό, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων εθνικών συστημάτων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προκλήσεις ε, των διασυνδέσεων για παράδειγμα ε, και κυρίως σε χώρες όπως η Ισπανία ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια της παροχής και να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα για τις ανανεώσιμες Επίσης, ποιος θα έχει την τελική ευθύνη ανάμεσα στις ε, ΤΕΣΕΟ και το επίπεδο το περιφερειακό. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόχλιτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Εγώ έχω δουλέψει στην βιομηχανία και πάντα είχαμε απόθεμα ή εν πάση περιπτώσει εναλλακτικέ πηγέ ενέργειας ε, για διάφορες ε, τεχνολογίες, ε, είτε ήταν κομπιούτερ, είτε οτιδήποτε τεχνολογία και αν ήταν. Αλλά πάντα είχαμε τέτοιου είδους ανακτικές πηγές παροχής ενέργειας. Τώρα συζητούμε το θέμα αυτό και νομίζω ότι το θέμα των, ε, του αποθέματος ε, είναι σημαντικό. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να αποθηκεύσουμε ε, ενέργεια, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε διπλές υποδομές, να έχουμε και μια δυνατότητα αντικατάστασης η οποία θα εξασφαλίζει σε, σε κάποιες περιπτώσεις την παροχή. Στην Ιταλία έγινε κάποια στιγμή ένα συνολικό blackout ακριβώς λόγω της έλλειψης αυτών των υποδομών, όπως και στην Πολωνία, όπως το είπε ο εισηγητής. Τι είναι λοιπόν σημαντικό, είναι σημαντικό να έχουμε εναλλακτικέ πηγές παροχής ενέργειας και τι εννοώ. Πηγές με βάση το φυσικό αέριο ή το νερό Αυτές είναι πηγές ενέργειας, τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως αποθεματικά. Νομίζω αυτές οι πτυχές είναι σημαντικές και μπορούμε να τις ενσωματώσουμε στην έκθεση. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι σημαντική και σε, κάποια, σε κάποιες χώρες υπάρχει και ε, συγκεκριμένο δικαίωμα των καταναλωτών να έχουν, να λαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια. Ευχαριστώ. Από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η κυρία Βερχέβεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ε, παρατηρήσεις τους, για τις προτάσεις τους ε, απέναντι στη δική μας πρόταση. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακούμε ότι γενικώ θεωρείται ότι είναι χρήσιμη η πρότασή μας ε, και απαντά σε μια ανάγκη να αντιμετωπίσουμε ένα νομικό κενό όταν υπάρχει όντως ανάγκη να συνεργαστούμε καλύτερα για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση κρίσεων. Και επίση μα ικανοποιεί το ότι θεωρείται ότι η πρότασή μα είναι ισόρροπη. βεβαίω, ακούμε και κάποια σχόλια που έχουν να κάνουν με τεχνικέ ανησυχίε, ανησυχίε ότι αφορά κάποιες λεπτομέρειες και Επίση, ε, κατανοώ και την ανάγκη που υπάρχει για περαιτέρω τεχνικέ συζητήσει Από τη δική μα την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί είμαστε πάντα έτοιμοι να σα παράσχουμε όλη την εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνική που έχουμε και να μπλακούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση που θεωρείται απαραίτητο να γίνει έτσι ώστε να προχωρήσει και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η πρόταση. Οπότε μπορείτε να βασίζεστε πάνω μα. Μια σύντομη παρέμβαση, ε, απάντηση. Καταρχά, ευχαριστώ ε, γιατί θεωρώ ότι η ε, πρόταση θα μπορέσει να βελτιώσει την παροχή ε, σε χαμηλό κόστος της ε, ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και όπως έχει υποθεί από τους ε, από τον εισηγητή και του Σκιώδη. Ε, είναι σημαντική η πρόταση αυτή ένα, και είναι σημαντικό κομμάτι του γενικότερου πακέτου γιατί έτσι θα εξασφαλίσει ότι οι αγορέ θα μπορέσουν να παραμείνουν ανοιχτές όσο δυνατόν περισσότερο ενώ εξασφαλίζουν ότι θα υπάρχει παροχή ηλεκτρική ενέργεια εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Ένα σύντομο σχόλιο για κάποια σημεία που ακούστηκαν και βεβαίω πάντα με την επιφύλαξη των ε, περαιτέρω τεχνικών συζητήσεων που μπορεί να χρειαστούν, ακούω κάποιε ανησυχίε για την ε, εμπιστευτικότητα των σχεδίων. Βεβαίω κατανοώ ότι κάποια ε, λεπτομέρειε των, των επιγόντων των σχεδίων πρέπει να είναι εμπιστευτικέ και δεν θέλω βεβαίω να δώσουμε οποιαδήποτε έμπνευση σε αυτού που θέλουν να κάνουν οποιαδήποτε επίθεση, αλλά στην πρότασή μα εμείς προβλέπουμε ότι θα υπάρχει εμπιστευτικότητα λέγοντας ότι μόνο τμήματα των σχεδίων αυτών θα είναι δημοσιεύσιμα. Οπότε ήδη προσπαθήσαμε να προβλέψουμε την ε, ύπαρξη εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Επίσης άκουσα κάποιες ανησυχίες ό,τι αφορά το διοικητικό άχθος. Να σας πω ότι το τελευταίο που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα αυξήσει το διοικητικό άχθος. Και γι' αυτό βασίζουμε την πρότασή μας ε, στα υπάρχοντα νομοθετικά πλαίσια. Δεν υποχρεώνουμε τα κράτη-μέρη να δημιουργήσουν νέα, νέες ε, δομές, νέες υποδομές. Ε, βασιζόμαστε σε αυτά που υπάρχουν ήδη και σε αυτά που ήδη έχουν δρομολογηθεί να υπάρξουν. Ε, περιφερειακά ας πούμε, επιχειρησιακά κέντρα που επίσης θα έχουν κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κρίσεων. Επίσης από πολλές πλευρές ε, ακούσαμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν σχέδια ετοιμότητας ό,τι αφορά του κινδύνου, αλλά και ε, αξιολόγηση και καταγραφή των κινδύνων για να ληφθούν ε, υπόψη οι διάφορες εθνικές ιδιαιτερότητες. Ως προς αυτό να πω ότι σε όλη μας την πρόταση, όταν εκπονούσαμε την κοινή μεθοδολογία, βεβαίω η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, προβλέψαμε να υπάρξουν και εθνικέ δυνατότητε αξιολόγηση. Οι εθνικέ αυτέ δυνατότητε αξιολόγηση υπάρχουν για να λαμβάνουν υπόψη του ακριβώ την εθνική κατάσταση. Υπάρχει περιφερειακή αξιολόγηση που συμπληρώνεται από την εθνική ε, αξιολόγηση όταν αυτή χρειάζεται για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητε του κάθε κράτου. Και ακριβώ επειδή επιτρέπουμε να, γίνουν, ε, να ληφθούν υπόψη οι εθνικέ ιδιαιτερότητε, τα εθνικά ε, σχέδια μπορούν επίσης να καλύψουν συγκεκριμένες εθνικές περιστάσεις. Κάθε χώρα είναι διαφορετική, έχουν διαφορετικά μείγματα ενέργειας και αντιμετωπίζει διαφορετικούς κινδύνους. Αν είσαι στην Ιταλία, ένας σεισμός είναι ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Στο Βέλγιο, ας πούμε, δεν είναι τόσο σημαντική η πιθανότητα σεισμού. Οπότε αυτό θεωρούμε ότι ήδη έχει ενσωματωθεί στην πρότασή μας. Επίσης, Άκουσα κάποια αιτήματα να ενταχθούν κάποια παραπάνω στοιχεία στην ε, εκθέση έτσι ώστε να είναι πιο λεπτομερείς, ας πούμε ε, προστατευόμενοι ε, καταναλωτές και ορισμός τους. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί γιατί βλέπουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών για το ποιο θεωρείται προστατευόμενος καταναλωτής. Γι' αυτό προτείνουμε μια πολύ μινιμαλιστική προσέγγιση, έναν πολύ μινιμαλιστικό ορισμό και ελάχιστη δυνατή εναρμόνιση, προστατευόμενοι δηλαδή καταναλωτέ είναι αυτοί που πρέπει να προστατευθούν λόγω, ε, από την πλευρά της ασφάλειας. Και χρειάζεται περισσότερη ε, διαφάνεια. Αλλά δεν θέλουμε να εναρμονίσουμε τον ορισμό αυτό, γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος, μια που υπάρχουν πολλές διαφορές στην Ευρώπη για να γίνει αυτό. Και επίση κάτι σημαντικό. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια. Δεν ορίζουμε ποια θα πρέπει να είναι αυτά τα μέτρα. Αυτό που προτείνει η πρόταση για την προετοιμασία για τους κινδύνους, ότι θα πρέπει να, δοθούν, να δοθεί προτεραιότητα στα, αγορά, στα μέτρα της αγοράς, με τα μέτρα που δεν βασίζονται στην αγορά να είναι η, εξαίρεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα ε, θα οριστούν από τους ε, λομπίστες, ε, από τις ομάδες πίεσης, επειδή δεν τα ορίζουμε εμείς. Το κράτος μέλος είναι αυτό που θα ορίσει τα μέτρα που θα περιλαμβάνουν τα σχέδιά του. Και οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν αυτή τη δράση μετά από μια συμπεριληπτική διαδικασία διαβούλευσης με τη συμμετοχή ενός ευρέως φάσματος εμπλεκόμενων φορέων και από τους καταναλωτές και από τη βιομηχανία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα είναι μια ομάδα μόνο πίεση η οποία θα ορίσει ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει το κάθε κράτο μέλο. Πρέπει να είναι α, μια ενσυνείδητη απόφαση αυτή που θα πάρει το κράτο μέλο με όλε τι απαραίτητε πληροφορίε. Και ένα τελευταίο σημείο ό,τι αφορά ε, το θέμα της ευθύνης, ε, το οποίο ανεφέρθη σε σχέση με την ε, ασφαλή της παροχής. Αυτή η πρόταση δεν αλλάζει εδώ πέρα την ισορροπία, απλώς ζητά πιο συντονισμένη προσέγγιση. Δεν αλλάζει όμως την ισορροπία που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ευθύνη. Αυτό που θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε είναι μια συντονισμένη προσέγγιση με περιφερειακές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, αφήνοντας όμως του ε, εμπλεκόμενου φορεί να, να κάνουν τη δουλειά όπως κάνουν τη δουλειά ήδη μέχρι τώρα. Αυτά ήταν τα αρχικά μου σχόλια και πάλι χαίρομαι πολύ που μπορώ να συμβάλλω στη συζήτηση και βεβαίως προσβλέπουμε και σε μελλοντικέ συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ακριβώς αυτό όπως το είπατε για την ασφάλεια της προμήθειας φυσικού αερίου κατά τον ορισμό μα. εμείς προτείναμε ένα ελάχιστο για την προστασία των καταναλωτών και εναρμόνιση σε όλη την Ευρώπη. Μία δυνατότητα δηλαδή για εναρμόνιση τέτοιου ορισμού. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να παρακαλέσω τον κύριο Ζανονάτο, τον εισηγητή μας, θα τον ρωτήσω λοιπόν αν θέλει να συνοψίσει την συζήτησή μας, να κάνει δηλαδή λίγες ακόμη παρατηρήσεις. Ναι, Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο γιατί οι συνάδελφοι και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν είπαν πράγματα που μου φαίνεται μπορούν να συγκλίνουν προς ε, μια λύση θετική. Ε, ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει καλή δουλειά. Είναι προφανές ότι προκύπτει το γεγονό. το θέμα δηλαδή του κινδύνου στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματο, διατρέχει για κάποια άλλα θέματα και αυτά ήδη αναφέρθηκαν και θα δούμε πώ θα είναι δυνατόν να τα λάβουμε υπόψη ωστόσο, στο πλαίσιο τη δερμοδιότητάς μα. Ευχαριστώ του όσου πήραν το λόγο και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα με πρωτοβουλίε ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ακριβώ τι συνίσταται ε, όλο, αυτή, αυτό το, το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Χρονοδιάγραμμα. 1-22 Ιουνίου εξέταση του σχεδίου έκθεσης. 29 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Τέλη Ιουνίου θα είμαστε. Εξέταση των τροπολογιών 25 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία στην Ήτρε 28 Νοεμβρίου. Έχουμε τώρα το πακέτο καθαρής ενέργειας. Πολύ σημαντικό κομμάτι της, των νομοθετικών μας προτάσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περνάμε στο σημείο 7. Ε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ε, η συγητής είναι ο συνάδελφος Μόρτεν Χέλβικ Πέτερσεν. Και αυτή η πρόταση αποτελεί κομμάτι του χειμερινού κοπακέτου και συνδέεται στενά με άλλους φακέλους αυτού του, της δέσμης. Ειδικά με αυτές που συνδέονται με την αναθεώρηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχο έχει να, να ε, εξυγχρονίσει το κανονισμό άσερα, ώστε να αντικατροπηδίζονται οι νέες αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού Η υπόφασή μας λοιπόν θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις νέες προτάσεις, πώς θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τις υπάρχουσες. Στόχος ε, είναι επίσης να αλλάξουν οι κανονισμοί που προβλέπουν αλλαγές στις κανόνες αγοράς και ε, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Κάποιοι κανόνες λοιπόν εκεί θα πρέπει να αλλάξουν και εμεί πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι. Ε, λοιπόν Μόρτεν Χέλβεκ Πέτρεσεν. Μπορείτε να πάρετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Υπάρχουν σημαντικά ωφέλη που προκύπτουν από την ύπαρξη μια πραγματικής ενιαία αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να υπάρξει αγορά χρειάζεται βέβαια και κάποιο επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης που να, δίνει, να, προσφέρει τις συνθήκες για να υπάρξει αγορά. Ο ρόλος λοιπόν της, ε, των ε, ρυθμιστικών αρχών ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις ρυθμίσεις εκείνες που επιτρέπουν ε, ε, από νοικοκυριά μέχρι καταναλωτές μέχρι επιχειρήσεις να έχουν επαρκές ηλεκτρικό ρεύμα και ιδίως ε, εν ώψη του μέλλοντος της αγοράς ενέργειας που θα βασίζεται όλο και περισσότερο στην συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο συντονισμό στον τομέα αυτό. Το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της ενιαίας αγοράς και να βελτιωθεί έτσι η χρήση των πηγών ενέργειας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πρόταση αυτή κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ως συνεργασία ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και θα ακούσω με προσοχή τις απόψεις των συναδέλφων μου. Θα αρχίσω πάντως ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της που αποτελεί αναθεώρηση. Δεν είναι εκ βάθρων ε, αναδιαρρύθμιση της ε, αγοράς ενέργειας. Άλλωστε και το όνομα αυτό, ΕΙΣΑ, είναι, σημαίνει Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Τώρα εδώ έχω τρία σημαντικά θέματα σήμερα που νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Πρώτα, οι αλλαγέ που γίνονται στη διαδικασία λήψη αποφάσεων μέσα στον ίδιο τον Οργανισμό Συνεργασία ρυθμιστικων Αρχών Ενέργεια, ιδίω για τη χρηματοδότηση και στελέχωση του οργανισμού. Και η περιφερειακή συνεργασία. Όσον αφορά τι αλλαγέ ε, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων των ρυθμιστικών αρχών ενεργέργεια, εδώ χρειάζεται να εξεταστεί προσχετικά η νέα πρόταση, Καθώ και άλλε ενδεχόμενε λύσει, Αν θέλουμε μια ενιαία αγορά που να λειτουργεί ορθά, χρειαζόμαστε έναν ισχυρό οργανισμό ρυθμιστικών αρχών ενέργεια που να μπορεί να ανταποκρίνεται στι ανάγκε. Ε, δηλαδή θα πρέπει να αποφύγουμε ε, τις, τα διέξοδα και είμαι διατεθειμένος να συζητήσω όλες τις προτάσεις που ενδέχεται να γίνουν για λύσεις. Δεύτερο ζήτημα όσον αφορά δηλαδή τις χρηματοδικές πηγές και την στελέχωση του Οργανισμού Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, που για την ώρα είναι πολύ περιορισμένες, πολύ μικρότερες από αυτές που απαιτούνται για να επιτρέψουν στον οργανισμό να αποκριθεί στα καθήκοντά του. Η χρηματοδότηση χρειάζεται να φτάσει σε ένα επαρκές επίπεδο. Τα έχουμε συζητήσει αυτά τα τελευταία χρόνια με τον οργανισμό αυτό. Έχουμε ένα πρόβλημα λοιπόν με τις χρηματοδοτικές πηγές του ΕΣΑ. Υπάρχουν διάφορες ιδέες για την αντιμετώπιση και η ιδέα επιβολής, επιβολής μάλλον τελών σε ορισμένους από τους μηχανισμούς από πλευράς του οργανισμού. Πάντως, η χρηματοδότηση είναι σημαντικό θέμα για τον Οργανισμό ε, Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Χρειάζεται να συνεργαστούν καλύτερα και τα λεγόμενα ROC που είναι οι περιφερειακές αρχές ενέργειας Αυτά δεν μπορούν να ρυθμιστούν σε εθνικό επίπεδο, μπορούν να ρυθμιστούν μόνο σε περιφερειακό επίπεδο, όπου ο οργανισμός συνεργασίας θα πρέπει να είναι η αρχή η οποία θα ασκεί την εποπτεία. Για να μπορέσει ο οργανισμός αυτός συνεργασίας να επιτελέσει το ρόλο αυτό, χρειάζεται να έχει τις ε, αναγκαίες εξουσίες για να ζητεί τι προφορίες που χρειάζεται για να μπορεί να εκτελεί το έργο εποπτείας. Το ίδιο η περιφερειακή αυτή συνεργασία θα προωθήσει την ενιαγορά με τη λήψη αποφάσεων για την πρόθεση του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Σημαντικό θέμα, το οποίο έχει σχέση και με τα άλλα, με τους άλλους φακέλους του πακέτου καθαρής ενέργειας, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να τα δούμε αυτά στο σύνολό τους και να δούμε και ποιες είναι οι περαιτέρω διακλαδώσεις και του νομοθετήματος αυτού με ε, τους άλλους φακέλους. Αναμένω μεγάλο ενδιαφέρον την συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους και τις συναδελφούς, ελπίζοντας ότι θα ε, μπορέσουμε να επιλέξουμε μια επικοδομητική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Λαϊκό κόμμα, ο κύριος Ρόιλ που είναι σκιώδης εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τις συζητήσεις που έχουμε διεξαραγεί μαζί του και για τις ιδέες του. Έρχομαι στα όσα είπε. Για να λειτουργήσει η νέα αγορά χρειαζόμαστε καλή συνεργασία και νομοθεσία. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι τα νομοθετικά εργαλεία που διαθέτουμε είναι επαρκή ή όχι. Αποδίδουν ή όχι. Και το ερώτημα που έχω θέσει σε όλους τους συνομιλητές μου ως τώρα είναι πού εντοπίζονται τα προβλήματα. Εν τέλει, έχω μονάχα δύο υποδείξεις. Αφενός ότι σε ορισμένα σημεία μεταξύ χωρών μελών υπάρχει το πρόβλημα ότι η εμπορική ε, συναλλαγή δεν λειτουργεί επαρκώς. Για παράδειγμα, Δανία, Γερμανία. Εδώ έχω ένα καλό παράδειγμα. Εάν εξετάσει κανείς πιο προσεκτικά τα πράγματα όμως θα δει ότι δεν είναι ζήτημα βελτιωμένης εποπτείας ή συνεργασίας, δεν λειτουργεί. Εφόσον σε ένα σημείο έρχεται πολύ ρεύμα, αλλά από την άλλη πλευρά των σύνορων δεν υπάρχουν επαρκείς αγωγοί για να διοχετευτεί περαιτέρω το ρεύμα αυτό, ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, εδώ δεν χρειάζεται περισσότερη συνεργασία ή βελτιωμένη συνεργασία, δεν χρειάζεται περισσότερα δίκτυα. Από την πλευρά τη Ομοσπονδιακή Γερμανία δεν έχουμε επαρκή δίκτυα. Άρα χρειαζόμαστε επέκταση δικτύων. Αυτό συμβαίνει συχνά. Λέμε χρειαζόμαστε περισσότερε αρμοδιότητε, καλύτερη οργάνωση κλπ. Όχι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει επαρκέ δίκτυο. Όσε αρμοδιότητε και να έχετε. Αν δεν έχετε δίκτυο, καμιά φορά επίση δεν γίνονται οι συμφωνίες αυτές επαρκώς γρήγορα, λένε ορισμένοι. Όμως, λένε ορισμένοι, δώστε περισσότερες αρμοδιότητες στους κεντρικούς οργανισμούς εποπτείας ή διαφορετικές προθεσμίες για να προωθηθούν, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Αυτό που ενοχλεί είναι ότι η απάντηση που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι χρειαζόμαστε ακόμα πιο ενισχυμένη, ακόμα πιο έντονη θεσμική συνεργασία και τότε θα λειτουργήσουν τα πράγματα. Αυτό δεν είναι αληθές. Δεν ισχύει. Το τρίτο τώρα. Αν θέλουμε να, να ε, αποδώσει συνεργασία, η ρύθμιση που έχουμε στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών με κάθε κράτος μέλος μία ψήφο και ενισχυμένες πλειοψηφίες, εγώ νομίζω δεν αποδίδει. Να υπάρξουν ενισχυμένες πλειοψηφίες, λέει άλλος, αυτό όμως δεν πρόκειται να αποδώσει. Γιατί πάμε να λύσουμε το πρόβλημα με τη βία. Δεν έχει νόημα να προωθούμε περισσότερες αρμοδιότητες στον κεντρικό οργανισμό, ενώ τα προβλήματα πρέπει να λύγονται στο περιφερειακό επίπεδο που πρέπει να γίνουν σχετικές προσαρμογές. Αυτό δεν μπορεί να το εποπτεύει ο κεντρικός οργανισμός. Προσοχή λοιπόν, όχι περισσότερες αρμοδιότητες των ΕΣΑ. Υπάρχουν ευφιέστερες λύσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Και αν ρωτήσετε ποια και πόσα προβλήματα υπήρξαν, πολλοί είναι οι περιπτώσεις που σας, ε, που σας αναφέρουν. Πολύ περιπτώσεις προβλημάτων. Τότε γιατί όλη αυτή η προσπάθεια λύσεων. Ούτως ή άλλως ο κόσμος αντιδρά αλλεργικά όταν λέμε ότι θέλουμε ντε και καλά να αυξήσουμε τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά πού αυτό είναι αναγκαίο και πού όχι. Εδώ δεν είναι αναγκαίο. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Πόχε των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ε, ευχαριστώ. Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. έχει τονίσει κατ' επανάληψη η Επιτροπή μας την ανάγκη επεκτάσεως των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για να παίξει τον ρόλο της στην αγορά ενέργειας. Αυξανόμενος ρόλος των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ο οποίος ασκεί μεγαλύτερη πίεση στον συντονισμό μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Η λεπτομερής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Συνεργασίας, αυτό είναι ένα στοιχείο που περιλαμβάνει τι προτάσεις τη Επιτροπής και το θεωρώ πολύ θετικό. Το ίδιο και η απλοποίηση των διαδικασιών λήψη αποφάσεων. Κατά τη γνώμη μου πάντως, εδώ υπάρχουν τρεις τομείς όπου θα πρέπει να εγκύψουμε στις συζητήσεις. Και πρώτο, η περιφερειακή συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και των διαχειριστών των δικτύων. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα συχνά υφίστανται την κριτική και όχι μόνο από αυτούς που διαχειρίζονται τα δίκτυα. Συχνά υφίστανται κριτική και από άλλες σκοπιές. Δεύτερο, με ενδιαφέρει η ανεξαρτησία του οργανισμού συνεργασίας. Η γνώμη μου είναι ότι ο οργανισμός συνεργασίας ρυθμιστικών αρχών ενέργειας πρέπει να είναι ελεύθερος από οποιοδήποτε πολιτικό δικτάτ, είτε από το εθνικό επίπεδο είτε από το ευρωπαϊκό. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε διαρκώς υπόψη μας. Τέλος, και αυτό νομίζω είναι και το πιο ακαθόδες ζήτημα, η χρηματοδότηση του Οργανισμού Συνεργασίας. Για να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία του ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο θα ήταν για ορισμένες δραστηριότητες του οργανισμού να μπορεί αυτός να επιβάλλει τέλη. Ισουαρές. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε, ο κύριος Χένκελ από την ομάδα ECR θα σα τα πω στα γερμανικά γιατί έχω μπροστά μου όλα τα έγγραφά μου στα γερμανικά ενώ συνήθως μιλώ τα αγγλικά. Πρώτα ορισμένες γενικότερες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι η ενιαία αγορά είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τώρα. Μπορεί να πει κανείς μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ενιαία αγορά δεν θα μπορούσε καν να υπάρχει. Δεύτερη προκατακτική παρατήρηση. Η Ενεργειακή Ένωση, η ενιαία αγορά ενέργειας δηλαδή, είναι σωστός στόχος και είναι σωστός στόχος για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία όμως αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα διότι αφενός θέλουμε να υπάρξει η ενιαία αγορά και για τα αγαθά και για τις υπηρεσίες και το καθεξής, αλλά την άλλη μεριά λέμε ότι κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να αποφασίζει η ίδια το μείγμα ενέργειας, το energy mix. Εδώ βρίσκεται μια εσωτερική αντίφαση, η οποία εμφανίζεται διαρκώς στις συζητήσεις αυτές. Τρίτο, στη συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνεται βεβαίως η αρχή της επικουρικότητας που εμείς ιδίως στη δική μου πολιτική ομάδα την επικαλούμαστε συχνά. Εξ τώρα όμως, εάν παραιτηθούμε από την αρχή της επικουρικότητας διότι θεωρούμε ότι γίνεται καλύτερα τα πράγματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα πρέπει να αποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όποιο άλλο ενδιαφέρεται ότι έχουν άδικο αυτοί οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στα παλαιά. Νομίζω πάντω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει κάποια θετικά επιχείρηματα για να αποδείξει αυτό που λέει. Δηλαδή ζητεί περισσότερα πράγματα. Θέλει να εξασφαλίσει όχι μόνο την προμήθεια, αλλά ζητάει και περισσότερο ανταγωνισμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πτυχή που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Με την ευκαιρία να μου επιτρέψετε να πω ότι εκθέσεις για ενδεχόμενο blackout τον Γενάρη στην κεντρική Ευρώπη έρχονται και πανέρχονται διαρκώς από ορισμένου που επικαλούνται ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα πράγματα στα χέρια των χωρών μελών μόνο. Υπάρχει όμως και το εξαντιθέτου επιχείρημα και τα λέει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν υπήρχε ένα σύστημα σαν αυτό που προτείνεται τώρα, πιθανότατα θα μειωνόταν σημαντικότατα ο κίνδυνος αυτός του blackout. Βεβαίως και χρειάζεται να συζητήσουμε ακόμη εάν η πρόταση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως συμβαδίζει με την αρχή της επικουρικότητας. Εμείς θα το κάνουμε αυτό και θα το προσέξει ιδιαίτερα η πολιτική μου ομάδα. Και εν τέλει να πω ακόμη ότι η ανεξαρτησία του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και η διαφάνεια των δράσεών του πρέπει να είναι απόλυτα εξασφαλισμένα. Διότι έχουμε και άλλες αρχές εποπτείας ή όργανα εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φροντίζουν για ελεύθερο ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να μπορέσει να είναι δυνατόν και στον τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τούρμες, ο οποίος αντικαριστά τον κύριο Σκέρλετς. Θα τα πω και εγώ στα γερμανικά, λέει ο κύριος Τούρμες. Ο κύριος Χένκελ έχει δίκιο που λέει ότι υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο εθνικό ε, μείγμα ενέργειας και στην ευρωπαϊκή προσέγγιση. Εγώ βλέπω μόνο μια διέξοδο, αφού δεν υπάρχει ούτως ή άλλως η δυνατότητα αναθεώρηση των συνθήκων για ιστορικούς λόγους. Να δούμε τι έχει νόημα οικονομικά. Σπάνια, σπάνια διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα από την Πορτογαλία στην Εστονία για παράδειγμα. Αλλά από την άλλη μεριά και η γερμανική αγορά ρεύματος δεν υπάρχει πλέον ούτε και η γαλλική. Διότι αν ήταν έτσι η Γαλλία, αν είχε μόνο εθνική αγορά ενέργεια δηλαδή, θα είχε πέσει blackout φέτο το χειμώνα. Ήρθε ρεύμα παλού. Υπάρχουν λοιπόν περιφερειακές αγορές ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν νόημα και οικονομικά. Με συνεργασία Γαλλίας, χωρών Μπενελούξ, Γερμανίας, Αυστρίας κλπ που οδήγησαν και σε πτώση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό το χρειαζόμαστε απαραίτητο και για την νοτιοανατολική Ευρώπη για να μπορέσει να υπάρξει και εκεί μια βελτιστοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Άρα χρειαζόμαστε περιφερειακές διασυνοριακές συνεργασίες, κάτι το οποίο έχει νόημα και οικονομικά αλλά και πολιτικά. Αν όμως καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, χρειαζόμαστε βεβαίως τότε και κάποιον ο οποίος θα διασφαλίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία δεν οδηγεί σε κατάτμιση των κανόνων. Δηλαδή, η ενιαία αγορά ανάμεσα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να έχει διαφορετικούς κανόνες από αυτούς που είναι στη Βόρεια Ευρώπη για παράδειγμα. Εκεί είναι ο ρόλος του ΕΣΑ. Αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν οι εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά χρειάζονται κάποιον ο οποίος να έχει τη συνολική αυτή επισκόπηση της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να τα καταφέρουμε, πρέπει να δώσουμε στον Οργανισμό συνεργασία Ρυθμιστικών Αρχών ενέργεια τις αναγκαίε αρμοδιότητε, την αναγκαία εποπτεία, χωρίς να τον φτάσουμε να γίνει ένας υπεροργανισμό. Αυτό είναι το καθήκον που έχουμε μπροστά μα. Ο Χέρμπερτ έχει δίκιο όταν λέει ότι αυτό που χρειάζεται, ο Χέρμπερτ δηλαδή, αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι η επέκταση των δικτύων. Όσο τα καλώδια περνούν από τον βορρά προς τον νότο, η Γερμανία δεν μπορεί να ανοίξει την αγορά της στη Δανία. Όσο υπάρχουν, για παράδειγμα, στο βορρά της Γερμανίας τα πάρκα αιωρικής ενέργειας. Αλλά χρειάζονται προθεσμίες Εάν όμως δεν επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται και κάποιος ο οποίος ως η ίστατη καταφυγή να μπορεί να λειτουργεί όταν δεν συνεννοούνται δύο ή τρεις χώρες περιφερειακά. Και εκεί βλέπω ένα ρόλο πάλι για τον Οργανισμό Συνεργασίας. Εάν δηλαδή μετά από την παρέλευση των προθεσμιών αυτών δεν εμφανίζονται ικανές οι εθνικές αρχές να συνεργαστούν. Χρειαζόμαστε βέβαια και μια ελάχιστη ροή πληροφοριών και ο οργανισμός χρειάζεται και κάποια χρηματοδότηση. Διότι οικονομικά δεν έχει νόημα να έχω μια αγορά συνολικής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων και να μην μπορώ να βρω κάποια λίγα εκατομμύρια για να εξασφαλίσω μια ρύθμιση η οποία θα ρυθμίζει τα, τα απαραίτητα. υπενθυμίζω ότι όταν καμιά φορά ξεσπά ένα σκάνδαλο insider trading, θυμάστε που είχε πριν από λίγα χρόνια γίνει κάτι τέτοιο, το αντιμετωπίζουμε. Και όμως δεν δίνουμε τα μέσα στον οργανισμό συνεργασίας για να αντιμετωπίσει τα πράγματα αυτά. Οικονομικά λοιπόν αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ε, επαναλαμβάνω μπορούμε να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια με την ενιαία αυτή αγορά. Αλλά Χρειαζόμαστε έναν οργανισμό συνεργασίας που να μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Όχι κανέναν υπεροργανισμό, αλλά ένα οργανισμό ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με κάποιον από τους πρώτους ομιλητές που λένε ότι δεν χρειαζόμαστε ενίσχυση της ε, υπηρεσίας η οποία θα, υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το παρόν έχει το συντονιστικό τους ρόλο. εξασφαλίζεται ο συντονισμός που μπορεί να παράσχει και αυτό υπάρχει και λειτουργεί. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να προτείνει πώς θα συνδεθούν τα δίκτυα μεταξύ τους, μεταξύ των διαφόρων χωρών. Όσο ισχυρή και αν είναι μία ε, υπηρεσία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να συνδέσει τα δικά μας ε, ε, δίκτυα, ας πούμε, τα δίκτυα της Αιχίας με την Πολωνία. αν τώρα κάνουμε μια νέα, δημιουργήσουμε μία νέα υπηρεσία η οποία θα προτείνει μόνο αυτό, ε, δεν ξέρω τι νόημα έχει. Ε, λοιπόν, το πράγμα το όπως έχουν είναι καλά, πιστεύω εγώ, η συνεργασία των υπηρεσιών λειτουργεί και όσο δεν έχουμε σωστή υποδομή, σωστά δίκτυα σε όλη την, Ευρώπη, δεν μπορούμε να δώσουμε νέες αρμοδιότητες σε αυτή την υπηρεσία. Γιατί δεν θα οδηγήσει σε τίποτα, δεν θα βοηθήσουν σε τίποτα αυτές οι νέες ε, αρμοδιότητες. Τώρα, για την, για την κατανομή των αρμοδιοτήτων, ναι, σωστά είναι αυτά που λέγονται στην πρόταση. Μπορούμε να το καταστήσουμε ακόμη πιο σαφέ για το πώ θα γίνεται η συνεργασία, η οποία μέχρι τώρα βεβαίω είναι πολύ επιτυχή. Πώ μπορεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Τα περιφερειακά κέντρα επίση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Μέχρι στιγμή έχουμε καταφέρει σε διημερέ επίπεδο να ε, διαρθρώσουμε τις σχέσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών με πολύ καλό τρόπο. Αυτό που δεν έχουμε επιτύχει είναι μετά την ε, ε, ένταξη της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας αυτό το κομμάτι του δικτύου να το συντονίσουμε. Αυτό όντως δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε. Και μέχρι στιγμής υπάρχουν, ε, έχουν περάσει 30 χρόνια από την επανένωση της Γερμανίας και ακόμη η Γερμανία ως μία χώρα δεν έχει ένα ενίο δίκτυο. Αλλά όσο ισχυρή και να είναι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να φανταζόμαστε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσίας. Τώρα, η χρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι έχει ρυθμιστεί πολύ καλά. Και δεν πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε χρηματοδότηση νέας υπηρεσίας, νέου φορέα, επειδή δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, για το ενεργειακό μείγμα. Ε, πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν. Το ενεργειακό μείγμα δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι πώς παράγω ενέργεια. Αν έχω αέρα, παράγω ε, ε, ενέργεια μέσω του αέρα. Αν έχω πολύ νερό στη χώρα μου, παράγω ενέργεια μέσω αυτού. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ήλιο αν έχω ηλιόλου, αν ζω στη χώρα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ε, επηρεάσει Κανένας. Καμιά υπηρεσία δεν μπορεί να επηρεάσει το πώ θα παράγεται η ενέργεια στη χώρα. Το ενεργειακό μείγμα αυτό που μας λέει είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ε, απαραίτητη ποσότητα παραγωγής, ε, παραγωγή μάλλον απαραίτητης ποσότητας ενέργειας. Α πούμε στη Βουλγαρία έχουμε πυρηνικού αντιδραστήρε. Χωρί να έχουμε εξασφαλίσει ότι η Βουλγαρία μετά το κλείσιμο αυτών των αντιδραστήρων μπορεί να έχει επαρκή παραγωγή ενέργειας. Ευχαριστώ. Και, πρόεδρος, ε, βεβαίως πρέπει να δούμε όντω πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τους πόρους μας. Εκ μέρου τη επιτροπή. έχουμε εκπρόσωπο της Γενικής ε, Διεύθυνσης Ενέργειας, τον κύριο, τον κύριο Φλόριαν Ερμακόρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μας το στοιχείο κλειδί είναι η αγορά ενέργειας να γίνει πιο αποτελεσματική. Και βλέπουμε ότι το βασικό θέμα εδώ είναι να έχουμε μια, ένα στενότερο συντονισμό για την, ε, μεταξύ των operators, των παρόχων, των ε, συστημάτων ε, παροχής. Αν γίνει αυτό και σε συνδυασμό με την καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο με τους παρόχους, θα έχει λιγότερο νόημα οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες να, να παραμείνουν στις εθνικές αρχές. Αλλά θα μπορούν να αποδοθούν αυτές οι αρμοδιότητες σε μια πλατφόρμα συνεργασίας. Αυτή, αυτό το ρόλο δηλαδή έχει να παίξει ο, ε, η υπηρεσία Acer. Οπότε χρειάζονται ναι, ε, νέοι πόροι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αρμοδιότητες, αλλά αυτό που κάνουμε εδώ είναι ουσιαστικά να προωθούμε την εσωτερική αγορά ενέργειας. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται πιο ε, ισχυρή εποπτεία από την πλευρά του Acer. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πάροχοι. Ε, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Δεν έχουν σημαντικό ρόλο μόνο οι ρυθμιστέ, ούτω ή άλλω οι υπηρεσίε είναι λίγο διαφορετικέ. Αυτό δεν το αρνείται κανεί. Αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν, ε, ένα σύστημα πλήρους ελέγχου, χωρίς όμως να υπερφορτώσουμε και να υπερρυθμίσουμε τα πράγματα. Ο συνάδελφος Πέτερσεν δεν ξέρω αν θέλει καταληκτικά να κάνει κάποια σχόλια. Ο εισηγητής, ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Κάποια από τα σημεία κλειδιά ήδη έχουν συζητηθεί όπως είπε ο κύριος Χένκελ πολύ σωστά, έχουμε αυτό το δίλημα. Από τη μία θέλουμε να έχουμε μια καλώς ενεργούσα αγορά, από την άλλη θα έχουμε, θέλουμε να εχουμε μια καλό ενεργουσα αγορα απο την αλλη θελουμε να εχουμε και το ενεργειακό μείγμα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε τη διατήρηση των ε, ωφελιών που μπορούμε να έχουμε από την εσωτερική αγορά ενέργειας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μελετήσουμε πιο προσεκτικά. Και βεβαίως υπάρχει ακόμη πολύ υλικό, πολλοί υπολογισμοί στις διάφορες αξιολογήσεις αντικτύπου που δείχνουν τα ωφέλη της ε, πιο ε, εντατικής συνεργασίας και συντονισμού. Βεβαίως πρέπει λοιπόν αυτό να το προσεγγίσουμε πιο προσεκτικά. Και επίσης συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ρόιλ για την επικουρικότητα. Αν υπάρχουν ωφέλη, το είναι η απόδειξη ακριβώς της ανάγκης του περαιτέρω συντονισμού και συνεργασίας και διασυνοριακά αλλά και περιφερειακά. Οπότε πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες συγγητές και βεβαίω προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μας για το φάκελο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης 10-11 Ιουλίου. Ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Κάποιους μήνες μετά, δύο μήνες μετά συγκεκριμένα, 6 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι. 6 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ε, ψηφοφορία στην Ήτρα 28 Νοεμβρίου και ψηφοφορία στην ε, Ολομέλεια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Οπότε κλείνουμε το σημείο. αυτό, θα το κλείσουμε το φάκελο αυτό τον Νοέμβριο ουσιαστικά. Σημείο 8. Feedback από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Ε, ασφάλεια παροχής αερίου και ο κανονισμός πρίμα. Να πω δύο πράγματα για την ασφάλεια της παροχής αερίου εγώ και τις διαπραγματεύσεις. Έγινε ένας τρίτος τριμερής διάλογος στις 27 Μαρτίου. Και ο τέταρτος προετοιμάζεται για την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμερούς διαλόγου, ο οποίος κράτησε 9 ώρες, οι διαπραγματεύσεις ε, προχώρησαν σημαντικά σε αρκετούς τομείς. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της αλληλεγγύης, το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε σωστά τους ε, προστατευόμενους ε, καταναλωτές, ορισμός επίσης του προστατευόμενου καταναλωτού. Η περιφερειακή συνεργασία, άλλο ένα σημαντικό θέμα, επί τη βάση των ε, διαδρόμων ε, επίγουσας παροχής ενέργειας. Εκεί είπαμε ότι χρειάζεται περισσότερη ε, ευελιξία. Υπήρχε αυτό βέβαια και στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και συμπερίληψη των μέτρων ενεργειακής επάρκειας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της παροχής αερίου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικό στο μέλλον. Έχουμε βεβαίως ένα σημαντικό πρόβλημα. οι κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών και τις κοινοποίηση. Οπότε προετοιμαζόμαστε σχετικά για τον τελευταίο τριμερή διάλογο που θα γίνει σε δύο μέρες. Είμαστε σε συνεχή επαφή, οι σκιώδες εισηγητές και βεβαίως ξέρουμε ότι και το Συμβούλιο ε, δουλεύει πολύ εντατικά πάνω στο θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι και αυτοί θα είναι έτοιμοι έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό τότε την εβδομάδα. Αλλά βεβαίως δεν μπορώ να προκαταλάβω οτιδήποτε. Οπότε Τετάρτη 26 Απριλίου θα διεξαχθεί ο τέταρτος τριμερής διάλογος. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις ή αν θέλετε να παρέμβετε. Ο κύριος Τούρμας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι επί της ουσίας. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω το Γέρζη και όλη την ομάδα του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ καλά οργανωμένες οι διαπραγματεύσεις. Είχαμε πολύ καλή στρατηγική και όντως προωθήσαμε τον φάκελο όσο δυνατόν ε, περισσότερο στις τελευταίες συζητήσεις. Θα είμαστε ενωμένοι και αυτή την εβδομάδα και είμαι αισιόδοξο ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το ένα εκκρεμέ θέμα είναι τι είδους και πόσο πολλές πληροφορίες χρειαζόμαστε από τις συμβάσεις έτσι ώστε να έχουμε μια καλή γενική εικόνα για, τον, για να προγραμματίσουμε την παροχή ασφάλειας σε περιπτώσεις επίγουσες. Αυτό λοιπόν το θέμα θα είναι αρκετά α, καυτό και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να κερδίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Η δική μας προσέγγιση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενιαία. Είμαστε πραγματικά ενωμένοι ως Κοινοβούλιο και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να διαπραγματευτεί κανείς με το Συμβούλιο. Το ίδιο έγινε και στι διαπραγματεύσει για το roaming, στο πακέτο για τη τηλεπικοινωνία. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλούσε με μία φωνή. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για μας να διαπραγματευτούμε. Και το ίδιο συμβαίνει και για την ασφάλεια της παροχής αερίου. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συζητητές, τις πολιτικές ομάδες, τους κοιόδες που ακολουθούν όλη την ίδια προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους πολίτες μας βεβαίως όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις, όχι μόνο για τους ε, προστατευόμενους καταναλωτές, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας και τη βιομηχανία. Αυτά έχω να σας πω εγώ για την ασφάλεια της παροχής αερίου. Επόμενο σημείο είναι ο κανονισμός πρίμα. Η κυρία Σακοράφα έχει το λόγο. Κατευθείαν από το αεροδρόμιο φαντάζομαι ήρθατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ. 11 Απριλίου οι, τα τρία θεσμικά όργανα συναντήθηκαν για τον τριμερή διάλογο, για το πρίμα. Και ξεκίνησαν οι συζητήσεις. Αλλά εντάξει, ας μην πω εγώ άλλα, γιατί μπορείτε να μας πείτε εσείς πολύ περισσότερα. Είναι δικό, δικό σας επίτευγμα αυτό και όλων των σχεδόν εισηγητών βεβαίως. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση να σας ενημερώσω ότι στις 11 Απριλίου του 2017 η διαπραγματευτική ομάδα της ΙΤΡΕ μαζί με την Μαλτέζικη Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διαργασίες του Τριλόγου για την υιοθέτηση της ευρωμεσαιρικής εταιρικής σχέσης πρίμα την πρώτη εταιρική σχέση με νομική βάση το άρθρο 185 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αυτή της Μεσογείου ενώ, όπως έχω τανίσει κατά επανάληψη, το πρίμα είναι μία από τις σπάνιες προσπάθειες επιστημονικής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκπατρισμού των κατοίκων της Μεσογείου και ταυτόχρονα φιλοδοξεί να προωθήσει στους τομείς των συστημάτων γεωργικών προϊόντων διατροφής και της διαχείρισης του νερού μια ολοκληρωμένη ενσωμάτωση σε επιστημονικό, διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο των χωρών στη Μεσόγειο. Τόσο προσωπικά υπό την ιδιότητα της εισηγήτριας και στο πλαίσιο της σχετικής εντολή της ΣΥΤΡΕ, όσο και οι συνάδελφοί μου σκιώδεις εισηγητές, προσπάθησαν σε εξαιρετικά ασφιχτικές χρονικέ προθεσμίε, να συμβάλλουν στη βελτίωση του νομοθετικού κειμένου, επικεντρώνοντας τη διαπραγματευτική μα προσπάθεια στη διασφάλιση του αμυγούς και αποκλειστικού πολιτικού χαρακτήρα των εφαρμογών και δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας, στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Διεθνέ Κοινοτικό Δίκαιο κατά την εφαρμογή του πρίμα, στην αναγνώριση του ανθρωπίνου δικαιώματο για πρόσβαση σε ασφαλέ, καθαρό, πόσιμο νερό και σε στοιχειώδει εγκαταστάσει αποχέτευση, στην ανάγκη το πρίμα να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών της περιοχής συμβάλλοντας στην βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας, της προστασίας και της βιωσιμότητα των συστημάτων γεωργικών προϊόντων διατροφής και της ολοκληρωμένης παροχής και διαχείρισης νερού, στην υποστήριξη από το πρίμα όλων των τύπων δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας για την πρόθεση έργων ενός ευρέως φάσματος τεχνολογικής ετοιμότητας και στην εξασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ μικρών και μεγάλων σχεδίων, στην ενίσχυση μια δίκαιη και ισορροπημένη γεωγραφική συνεργασία στο πλαίσιο τη ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, στην αποτροπή μια κατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών λαθρεπιβατών με την θέση συγκεκριμένων προποθέσεων και επαρκών δεσμεύσεων, στην ενδυνάμωση του ανοιχτού χαρακτήρα του πρίμα για όσε χώρε θέλουν να συμμετέχουν εφόσον τηρούν τι προποθέσει και στην εξασφάλιση διαφανού και αποτελεσματική διακυβέρνηση, διαχείριση και εφαρμογή του πρίμα. Και τέλος, και σε σχέση με την οριστικοποίηση του τελικού ύψους της κοινωνικής συνεισφοράς, σας ενημερώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι λόγω της αυξημένης δημοφιλίας του πρίμα, Τέσσερις επιπλέον χώρες και συγκεκριμένα η Κροατία, η Σλοβενία, η Αλγερία και η Τουρκία δήλωσαν πρόσφατα τη δούλησή τους να συμμετάσχουν με αποτέλεσμα να έχουμε 18 συνελικά χώρες να διεκδικούν μερίδιο από αυτή την πρωτοβουλία και ταυτόχρονα η Αίγυπτος και η Πορτογαλία που ήδη συμμετέχουν ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για αύξηση της συμμετοχής τους. Λαμβάνοντα υπόψη παραπάνω εξελίξει, η διαπραγματευτική ομάδα τη ΣΥΔΑ συμφώνησε στην αύξηση τη κοινοτική συνεισφορά στα 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται στα 220 εκατομμύρια ευρώ, η οποία κρίθηκε αναγκαία για την αποτελεσματική συμμετοχή των νέων κρατών, αλλά και λελογισμένη ώστε να μην διαταραχθεί σημαντικά εκ νέου η ισορροπία του, στην κατανομή του προγράμματο Ορίζοντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι όντα στην τελική φάση του νομοθετικού μα έργου, θέλω να εκφράσω ειλικρινεί ευχαριστίε ε, για την υποδειγματική συνεργασία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και ειδικά στη Μαλτέζικη Προεδρία που έθεσε το πρίμα ω πρώτη προτεραιότητα στον τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία, σε εσά κύριε Πρόεδρε, στου σκιώδει συζητητέ, στου συμβούλου των πολιτικών ομάδων, στου διαπιστευμένου βοηθού και στην γραμματεία τη ΣΥΤΡΕ. Ευελπιστώ στην γρήγορη και αίσια ολοκλήρωση των εργασιών μα με την υπερψήφιση του κειμένου στην επόμενη συνεδρία στη ΣΥΤΡΕ και κατόπιν στην Ολομέλεια του Ιουνίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθούν εγκαίρω οι ενδοενωσιακέ ενέργειε και η σύναψη των διεθνών συμφωνιών με όσε χώρε απαιτείται. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στο πρίμα να επιτευχθεί ο συλλογικό διοργανικό στόχο, να τεθεί δηλαδή το πρίμα σε πλήρη λειτουργία, επιχειρησιακή εφαρμογή από την 1η πρώτη του 2018, όπω όλε και όλοι επιθυμούμε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, thank you very much. Any other request for floor? Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ και εσάς ως εισηγήτρια και τους και οδησυγητές για την θαυμάσια συνεργασία. Πραγματικά ήταν μια ταχύτατη προσέγγιση από την πλευρά της Επιτροπής μας με θαυμάσια αποτελέσματα. με αποτέλεσμα ένα εξαίρετο νομοθετικό έργο. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν όλων των σχεδόν εισηγητών και της εισηγητρίας βεβαίως. Αύριο λοιπόν το πρωί στις 9 συντονιστές στις 10 προβλέπονται ψηφοφορίες. Υπενθυμίζω 10 η ώρα ψηφοφορίες στην ίδια αίθουσα που είμαστε τώρα. See you